Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών αιτήματα για τροποποιήσει στη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι διορισμοί αυτοί θα καταγραφούν στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης. Αν δεν προβληθούν ενστάσεις μέχρι την έγκριση των εν πρακτικών, οι διορισμοί αυτοί θα θεωρηθούν εγκριθέντες. Και τώρα περνούμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια